μας και πιο επίσημα. Ξεκινούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Right. Um, I'd like to... Uh, θα ήθελα... First of I'd like to... Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στη σημερινή συνεδρίαση. Ένα Καλώς ορίσατε και σε αυτούς που μας παρακολουθούν ζωντανά στο διαδίκτυο. Ε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Βγάλαμε μια ομαδική φωτογραφία η οποία σίγουρα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα μπορέσετε να μας δείτε όλους μαζί. Χαίρομαι πολύ που καταφέραμε να βγούμε όλοι μαζί αυτήν τη φωτογραφία. Ας προχωρήσουμε τώρα στη σημερινή μας δουλειά θα είναι μια πολύ άσχολη ημέρα ψηφοφορίας. Ε, πιστεύω πως είστε καλά προετοιμασμένοι. Αλλά πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, σήμερα το πρωί έχουμε την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, που είναι η κύρια ψηφοφορία μας. Θα ήθελα ο εισηγητής να μας την παρουσιάσει με λίγα λεπτά. Ε, έχουμε σημαντική δουλειά να κάνουμε, να εγκρίνουμε επίσημα τη συμφωνία που επετεύχθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση, αποτέλεσμα των του, επίσημου, του επίσημου τριμερούς διαλόγου. Υπάρχουν τρεις σημαντικοί φάκελοι. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών των καταναλωτικών διαφορών και η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Δυστυχώ η κυρία Τούν δεν κατάφερε να έρθει σήμερα. Νομίζω ότι ο κύριος Σβάμπ θα το παρουσιάσει στη θέση της. Καταρχήν θα ήθελα ε, ο Λουίς Γκρέκ που είναι ο εισηγητής ε, για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και αντιπρόεδρος της ομάδας μας να την παρουσιάσει. Έχω εδώ την επίσημη επιστολή από το Συμβούλιο, ε, έτσι μοιάζει, αυτή είναι, που λέει ότι το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι εάν υιοθετήσουμε αυτή τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση, που είναι η θέση της διαπραγμάτευσης, που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις, τότε το Συμβούλιο θα εγκρίνει την ε, έκθεση αυτή. Αυτό είναι τμήμα των ε, συμφωνιών μας για τη διαφάνεια. Όποιος θέλει να δει τις λεπτομέρειες μπορεί να τις βρει στην ιστοσελίδα μας. Ε, Λουίς Γκρέχ, θέλεις να πεις λίγα λόγια για τη συμφωνία. Και μετά ο Άντριου Σβάμπ και μετά έχουμε τον την εκπρόσωπο της Επιτροπής που και εκείνη θα πει λίγα λόγια. Λοιπόν, Λουίς Γκρέκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από την επιτυχή κατάληξη του τριμερούς διαλόγου στις 5 Δεκεμβρίου και την έγκριση του Κόπερμερ για, για το νομοθετικό κείμενο, μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές, σας ζητούμε να εγκρίνετε, να στηρίξετε το κείμενο. Ε, με μία εξαίρεση. Ε, που υιοθετήθηκε με βάση τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Νομίζω συνεργαστήκαμε πολύ καλά μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και καταλήξαμε σε μια ισορροπημένη ε, και δίκαιη έκθεση. Ωστόσο υπάρχει ένα μόνο σημείο όπως ανέφερα το οποίο θέλω να αναφέρω. Μία φράση συγκεκριμένα ε, στην αιτιολογική σκέψη 19 που λέει ή για δικαιολογημένους λόγους Νομίζω ότι η διατύπωση χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση. Θα την αποστείλουμε πίσω ε, στη νομική μας υπηρεσία και στους γλωσσολόγους μας ε, για να οριστικοποιήσουν ε, την διατύπωση έτσι ώστε να είναι σαφής και συνεπής με τη διατύπωση του υπόλοιπου άρθρου. Πέρα από αυτό έχουμε καταλήξει σε μια πολύ καλή συμφωνία. Νομίζω ότι οι καταναλωτές έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή την νομοθετική πρόταση. Ε, πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τον Hans Peter, τη Heider, τον, Robert, τον Robert Rochefort, καθώς και τον κύριο Ντέονγκ, τον κύριο Μπουζόη, που ήταν εισηγητής ε, από τη νομική πλευρά, και τον κύριο Φόξ. Χωρίς ε, την στήριξη και την ε, συνεργασία τους δεν θα βρισκόμασταν εδώ σήμερα. Είναι μία από τις λίγες εκθέσεις που έτσι προχωρούν με την πρώτη ανάγνωση, που, είναι έτσι, που έχουν τόσο καλή διάρθρωση και όλη η, εργασία, η όλη εργασία έγινε πολύ αποτελεσματικά. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή της καθώς και το Συμβούλιο. Πέραν τούτου, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, ε, για τον τρόπο που ηγήθηκες αυτής της προσπάθειας. Νομίζω σου, αξίζουν, σου αξίζει ένα χειροκρότημα. Άντριο Σβάμπ, θα πείτε λίγα λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να πω και τόσα πολλά στο στάδιο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που φτάσαμε εδώ και φυσικά ευχαριστώ και όσους δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα. Εντάξει λοιπόν, ε, θα ήθελα να ψηφίσουμε μαζί τις δύο αυτές εκθέσεις. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να κρατήσουμε και τα αρχεία μας. Άρχεται η ψηφοφορία έγκριση της, προτα... της πρότασης που έχουμε μπροστά μας ως αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Έχουμε 38 ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Παρακαλώ ψηφίστε όλοι. Ελέγξτε τις κάρτες σας, αν λειτουργούν, αν όχι. 39 έχουμε. Το σύστημα θα μας πει... Α, 40. 40 λοιπόν κάρτες και ένα άτομο δεν έχει ψηφίσει. Εμφανίζονται όλες οι κάρτες. Οι, σοσιαλ δημοκράτες έχουν ψηφίσει παραπάνω κατά μία ψήφο. Δεν είναι και τόσο σημαντικό σε αυτό το στάδιο. Περατούται η ψηφοφορία. 35 υπέρ, 4 κατά. Έχει λοιπόν εγκριθεί πανηγυρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι η κυρία Ρουσό να κάνει ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΜΚΟ για το σκληρό και πολύτιμο έργο τους, τους εισηγητές, την κυρία Τούν, τον κύριο Γκρέτ και όλους τους σκιώδεις ε, εισηγητές. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια καλή, ισορροπημένη συμβιβαστική λύση και τα τρία όργανα κατάφεραν να συμμορφωθούν και να υπηρετήσουν ε, τις πολιτικές υποχρεώσεις της εσωτερικής ε, Αγορά και να καταλήξουν σε συμφωνία το 2012. Είναι σημαντική πρόοδο για του καταναλωτέ για την εσωτερική αγορά, για την ανάπτυξη τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και καλά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τρόπο που εργαστήκατε με το... και με το Συμβούλιο. Πραγματικά υπάρχει και η πράξη της ε, ενιαίας αγοράς και έχουμε υπηρετήσει τις δεσμεύσεις μας και πάνω σε αυτό. Θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο που θα μας απασχολήσει όλο το πρωί. Εάν χρειαστούμε κάποιο διάλειμμα για καφέ θα σταματήσουμε. Εξαρτάται αν θα έχουν κουραστεί τα δάχτυλά σας από το να ψηφίζετε. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή να πει δύο λόγια και νομίζω ότι και ο κύριο Σβάμπ εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και ο κύριο Έγκελ θα θέλουν να πούν κάποια πράγματα και ίσω και οι άλλοι σκιώδει εισηγητέ πριν ψηφίσουμε. Κύριε Ταραμπέλα. Πρώτα εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για το τεράστιο έργο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πάει ένας, ένας χρόνος σχεδόν από τότε που η Επιτροπή πρότεινε αυτή την οδηγία πάνω στην οποία εργαστήκαμε επιτυχημένα, τηρήσαμε τις προθεσμίες, εργαστήκαμε σκληρά Ευχαριστώ τους σκιώδεις ε, εισηρητές Κρόιτσμαν, Ούλε, Χάρμπορ, ε, ε, τον κύριο Κορνελής Ντεγιόγκ, τον κύριο Σαλβίνη. Ευχαριστώ το προσωπικό μας, τη γραμματεία της Επιτροπής, η οποία εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά. Και έτσι καταφέρουμε να ψηφίσουμε σήμερα χωρίς να διακόψουμε για καφέ. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο. Καταφέραμε να έχουμε τις συμβιβαστικές μας τροπολογίες, ε, οι οποίες χαίρουν ευρείας υποστήριξης, όχι από όλες τις πολιτικές ομάδες προφανώς, γιατί και το αντικείμενο είναι στρατηγικής φύσεως και κατανοεί κανείς ότι υπάρχουν αποκλήσεις απόψεων πάνω σε ορισμένα από τα θέματα, από τα σημαντικά θέματα. Εκείνο που θελήσαμε ήταν προφανώς να οργανώσουμε καλύτερα τα δημόσια οικονομικά, ε, υιοθετώντα και προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία χαιρετώ, ευχαριστώ. Η στάση τη ήταν πολύ επικοδομητική σε όλε τι συναντήσει, συμμετείχε, ε, μα βοήθησε, μα καθοδήγησε και θα το πω και σήμερα. Ε, είχαμε την τύχη να εργαστούμε πάνω σε μια θετική πρόταση της Επιτροπής, πράγμα που δεν ισχύει τίποτα και το ξαναλέω εδώ, το έχω επαναλάβει πολλές φορές, γίνομαι και ενοχλητικός, αλλά πραγματικά ήταν πολύ καλό. Ε, και έτσι τώρα όλος ο κρατικός τομέας, κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση έχουν τώρα ένα μπούσουλα για το πώς θα οργανώσουν τα οικονομικά τους, ε, που θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που θα πληρούν και τους περιβαλλοντικούς όρους, τους κοινωνικούς όρους. Ε, επίσης θα επιλέγεται η οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά ε, επιλέγοντας ε, τους υπεργολάβους πάρα πολύ προσεκτικά, επιτρέποντας τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε έτσι ένα σωστό πλαίσιο που θα αποφεύγει την ε, διασπάθηση των δημόσιων πόρων και θα βοηθήσει τον κάθε συμμετέχοντα. Δεν θα μακρηγορήσω, δεν θέλω, έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη διαδικασία. Πάντως ευχαριστώ για την εργασία. Ήταν μια καλή εργασία, στέλνει ένα σωστό μήνυμα από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έδωσαν το χρόνο τους, που συμμετείχαν σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, που απαντούσαν στις επιστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανταλλάξαμε πάρα πολλές επιστολές μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το έργο και ως σκιώδης εισηγητής πραγματικά ξέρω ότι ήταν ένα τεράστιο έργο αυτό. Τώρα όμως πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Frank Angle; Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, ε, να ξεκινήσω με αυτό που πρέπει, με τα πρέποντα, δηλαδή να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή, τον Μάρκ Ταραμπέλα, καθώς και όλους τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές, για όλη τη δουλειά που κάναμε μαζί. Δεν ήταν και μικρό πράγμα, έναν ολόκληρο χρόνο διήρκησε για να ε, επιτύχουμε ε, και στο μέλλον, ε, να ξέρουμε ότι δεν τελειώνουν όλα εδώ, έχουμε και συνέχεια. Τα αποτελέσματα ίσως δεν είναι τέλεια και δεν αποκλείω μετά την ψηφοφορία να πρέπει να επανέλθουμε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια πάνω σε ορισμένα σημεία ε, και να το μαζέψουμε και να το φροντίσουμε κι άλλο το κείμενο. Εγώ συνεχώς ανακαλύπτω θέματα ε, και πολλές φορές πέφτω πάνω σε διατυπώσεις που δεν είναι υπρέπουσες. Η κυρία Άννα Μαλία Κοράτσα Μπίλντ, η συνάδελφος, θα προτείνει τρεις τροπολογίες προφορικές πριν από την ψηφοφορία. Θα δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Και στους, προς τους συναδέλφους μου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρέπει να τους πω ότι στην λίστα ψηφοφορίας θα πρέπει να δούνε την τροπολογία 253 η οποία ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θα δούμε λίγο και τις άλλες πολιτικές ομάδες, ο κύριος Μάντες, εκ μέρους της κυρίας Κρόιτσμαν, που θα έρθει λίγο αργότερα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους σκιώδεις εισηγητέ, τον κύριο εισηγητή και όλους όσους συμμετείχαν, γιατί ήταν τρομακτικό το έργο, πραγματικά και αυτό που είπε τώρα ο Φρανκ Άγκο στον ρόλο μου συντονιστή. Είναι δυνατό. Μήπως μετά από το αποτέλεσμα να κάνουμε μια αξιολόγηση πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, γιατί αυτό το νομοθετικό κείμενο αφορά την οικονομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τον κάθε πολιτικό της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, της κεντρικής κυβέρνησης, του ευρω... στο ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η νομοθεσία. Πρέπει να ψηφίζουμε νομοθεσία που να είναι εφαρμόσιμη. Υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα για την πρώτη πρόταση για τις δημόσιες συμβάσεις. Τώρα προσπαθήσαμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια ε, ή δυνατόν και αν μπορεί να συμφωνήσει ο εισηγητής να κάνουμε μια αξιολόγηση πριν περάσουμε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Να πραγματικά για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό ε, επιφέρει μια βελτίωση στην νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστώ κυρία Βουλέ. Θα είμαι σύντομη και εγώ νομίζω όπως είπε και ο Έγγελ ότι πριν από την Ολομέλεια πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του κειμένου θα πρότεινα οι συντονιστές να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη γι' αυτό, ούτω ώστε όλες οι ομάδες να συμμετάσχουν. Είναι σημαντικό πιστεύω αυτό και το λέω αυτό, σύμφωνο και με τους άλλους που το είπαν, ότι έχει μεγάλη σημασία η χορήγηση δημοσίων συμβάσεων. Αυτό που ψηφίζουμε σε όλα του τα σημεία πρέπει να έχει τη σωστή σημασία και την σωστή σαφήνεια. Πρόεδρος, να κλείσω εγώ ίσως την συζήτηση ως πρόεδρος. Α, α, με συγχωρείτε, κάποιον ξέχασα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ εσείς πρώτα και μετά εγώ. Ως κοιόδης και ως πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ήθελα να σας προσπεράσω, αλλά να το πω παρόλα αυτά. Υποστηρίζω τους προηγούμενους επανειλημμένα είπαμε να μελετήσουμε το θέμα αυτό πριν περάσουμε στην Ολομέλεια, τουλάχιστον από πλευρά των μικρομεσαίων, γιατί για αυτές είναι πολύ σημαντικό, καθώς και για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το κείμενο πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό. Αξίζει όντω λοιπόν την προσπάθεια. Ποτέ δεν ξέρουμε μετά από τόσε τροπολογίε. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε τι κείμενο θα προκύψει. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι παίρνουμε το θέμα αυτό στα σοβαρά Οπωσδήποτε συμφωνώ ότι είναι καλό να το συζητήσουν και να αποφασίσουν οι συντονιστέ. Είμαι ιδιαίτερο υπέρ αυτή τη ιδέα. Πρόεδρο. Συνολικά, το κείμενο αυτό ήταν πολύ περίπλοκο και νομίζω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή είναι πάντα μια ενδιάμεση φάση. Θυμόσαστε τι είπαμε για την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες που ήταν ε, το προηγούμενο μεγάλης έκτασης ε, νομοθέτημα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί. Εγώ δεν ήμουν τότε πρόεδρος, αλλά είχαμε πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Γιατί και πολλές άλλες επιτροπές έχουν εμπλακεί. Το κείμενο το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά εκείνη τη φορά με τις ε, υπηρεσίες και το βελτιώσαμε σημαντικά. Και έτσι είχαμε και ισχυρή στήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτή λοιπόν θα είναι η επόμενη φάση της διαδικασίας. Όσο καλά και αν το εκπονήσει ο εισηγητή με ένα τόσο περίπλοκο κείμενο, ορισμένα πράγματα θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Και στην ε, φίλη μου Κράτσα Μπέλτ, ε, να υποβάλουμε τώρα τροπολογίες σε αυτή τη φάση ε, δεν θα βοηθήσει. Μπορείτε φυσικά να το κάνετε, αλλά θα πρέπει να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο από όλες τις πολιτικές ομάδε για να μπορέσουν να υποβληθούν αυτέ τι τροπολογίε. Ε, αν επιμένετε εντάξει αλλά δεν το ενθαρρύνω αναγκαία ως πρόεδρος. Εδώ λοιπόν είμαστε. Τώρα πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Μετά θα δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Συμφωνώ και με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι δηλαδή τα βασικά στοιχεία αυτής της μεταρρύθμισης πρέπει να διατηρηθούν. Προσπάθεια απλούστευσης, προσπάθεια καλύτερης εφαρμογής και επίσης ε, πιο προσβάσιμο πρέπει να είναι αυτό το κείμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα ξαναβρούμε στην τελική μας θέση. Είναι βασικό σημείο. Ακόμη μπορεί να μην το έχουμε επιτύχει. Και οι συνάδελφοι που θέλουν να ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν, αλλά να το κάνουν ούτως ώστε να είναι αποδεκτό από όλους, για να μπορέσει μετά να είναι εφαρμόσιμο το κείμενο. Αλλά έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι με τις δυνατότητες που είχαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτή τη φάση το προσωπικό μας ε, όλους που είναι εδώ παρόντες αλλά και όλους τους βοηθούς των βουλευτών ήταν πολύ σημαντική εργασία ήταν ε, επική αυτή η προσπάθεια πριν από ένα χρόνο ακριβώς μας ε, εστάλει το κείμενο ο κύριος Φαμπ θέλει κάτι να πει. Με συγχωρείτε, συνήθως είμαι πολύ σύντομος. Αλλά θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Από πλευράς ΕΛΚ να διευκρινίσω το εξής. Σε πολλά σημεία δεχθήκαμε συμβιβασμούς που δεν ήταν εύκολο να περάσουν στην ομάδα μας. Το κάναμε αυτό ελπίζοντας, έχοντας κάθε εμπιστοσύνη και ελπίδα ότι έτσι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ευρεία συνένεση. Εάν όμως αυτή η συνένεση τώρα δεν είναι δυνατή, τότε αυτή η καλή θέληση που επιδείξαμε στις περαιτέρω ψηφοφορίες θα πρέπει να περιοριστεί. Ελπίζω λοιπόν οι συμβασμοί που έχουμε μπροστά μας, στα σημεία τα οποία ανέφερε ο ισκιώδης μας Έγγελ, μπορεί να υπάρξουν κάποιες ε, φραστικές βελτιώσεις, αλλά τελικά, τελικά θέλουμε να υπάρξει πολύ ευρεία συνένεση. Αυτό είναι ο στόχος μας για την τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευρά της ομάδας μου να διευκρινίσω απόλυτα ότι και εμείς κάναμε πολλές ε, παραχωρήσεις για να επιδιώξουμε και να επιτύχουμε συμβασμούς με τις άλλες ομάδες. Γι' αυτό με εκνευρίζει κάπως αυτό που ήδη άκουσα, ότι τώρα πρέπει να γίνει ένα νέο καθάρισμα του κειμένου. Καταλήξαμε σε τροπολογίες με όλες τις ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι εσωτερικά η ομάδα, οι διάφορες ομάδες, οι πολιτικές ομάδες συζήτησαν το θέμα αυτό. Στην ομάδα μου το κάναμε. Και νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν εκ των υστέρων μέσω της σημερινή διαδικασίας και επαναλαμβάνω και εγώ ότι θέλουμε ευρία πλειοψηφία ούτω ώστε να, αυτό που επιτύχαμε να μην ανατραπεί μετά στην Ολομέλεια. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καλό για την περαιτέρω συνεργασία στην Επιτροπή μας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε όντως προσεκτικοί. Όλες οι πλευρές έδωσαν και έλαβαν, να το πω έτσι. Δεν ήταν απλή η επίτευξη αυτών των τροπολογιών. Να μην προκύπτουν λοιπόν τώρα αμφιβολίες ότι όλα αυτά είναι προσωρινά, ότι οι συμφωνίες που καταλήξαμε ήταν παροδικές, το ζήτημα είναι και στην Ολομέλεια να καταλήξουμε σε τέτοιε θετικέ συνενέσει. Πρόεδρο, μα δεν νομίζω ότι το είπε κανεί κάτι τέτοιο. Αλλά θα δούμε τι θα προκύψει. Αλλά η φύση των συμβασμών είναι ότι πρέπει όλοι να δώσουν και να λάβουν. Να υπάρξει ντούνε και λαβίν. Λοιπόν, αν συμφωνείτε, να ψηφίσουμε τι συμβαστικέ τροπολογίε 65 και 83. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 66 όπου θα έχουμε κατά τμήματα κατά τέσσερα τμήματα λοιπόν ψηφοφορία υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται τρίτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία για το τμήμα 3 Κοιτάξτε, αργείτε πολύ να ψηφίσετε. Είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρέπει να προχωρήσουμε, αλλιώ δεν θα τελειώσουμε. Βλέπω μόνο 35 να έχουν ψηφίσει. Ε, τέσσερα άτομα έχουν βάλει τι κάρτε του στη σχισμή, αλλά δεν έχουν ψηφίσει. Παρακαλώ, ψηφίστε. Α, 39, ωραία. Παρακαλώ να ψηφίσετε πιο γρήγορα. Πέρα. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 24 κατά. Τέταρτο τμήμα. Τέταρτο υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Να περάσουμε τώρα στην 453 της κυρίας Ζούλα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Κατόπιν μαζί από κοινού για αυτές τις ψηφοφορίες που βλέπετε κατά απορρίπτονται. 650 δεν θα ψηφιστεί, έχει αποσυρθεί. 371 και 54. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Και τώρα έχουμε τρει τη κυρία Πετικά είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συμβαστική 74. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 80 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 67 υπέρ κατά εγκρίνεται οπότε περνάμε 407-408 θα πρέπει να τις έχετε αυτές υπέρ κατά απορρίπτονται 409 υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 409. Α, δεν ήταν ε, χωρί τη ψηφοφορία. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Δεν ήταν συγγνώμη από κοινού ψηφοφορία. Βάλαμε δύο μαζί να ψηφίσουμε την 408. Η πρώτη ψηφοφορία ήταν την 407. Τώρα είμαστε υπέρ 408. Ψηφίζουμε υπέρ κατά, απορρίπτει 408. Περνάμε στην 409. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία 409. Ψηφίσατε 40. Ε, ψηφίζουν 40, παρακαλώ γρήγορα. Μόνο 39. Δεν ξέρω ποιο είναι ο 400. Ωραία, εγκρίνεται. 27-11. 410. Υπέρ. Θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 410. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε πιο γρήγορα. Δεν βλέπω να προλαβαίνει το σύστημα. Το ηλεκτρονικό. Λοιπόν, 37, πέρας, πέρας. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Απορρίπτεται. Η 17 καταπίπτει, εφόσον εγκρίθηκε η προηγούμενη. Ρέτζι 26, ως προστήκη. Άρχεται. 26, προστίκη. Η ΕΛΚ, ψηφίζει ένα παραπάνω. Κάποιο να βγάλει την κάρτα του. Α, ωραία, ωραία. 39, πέρα. Εγκρίνεται. 21-18. Τώρα θα ψηφίσουμε από κοινού ταυτόσιμε τροπολογίες για το άρθρο 6. Ποιοι είναι υπέρ. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτονται. Ρέζι 27. Άρχεται Ρέζι 27. Πέρας. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην 68 συμβαστική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Μετά έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες εξαίρεσης. Ε, έχουμε εδώ από κοινού ορισμένες ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συγγνώμη, δεν ήταν πολύ σαφές. Αυτό το τμήμα μαζί, υπέρ, κατά, απορρίπτονται νομίζω. Νομική 14, ζουρί 14, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Είναι τα 18, Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Είναι τα 19. Άρχεται. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται. Συμβαστικέ 70 70-72 από κοινού αλλά κατά τμήματα βλέπετε που είναι το πρώτο και το δεύτερο τμήμα πρώτα απ' όλα το κύριο κείμενο υπέρ κατά εγκρίνεται και μετά το τμήμα 2 με την προσθήκη αυτών των λέξεων άρχεται η ψήφιση αυτών για το δεύτερο τμήμα της τμήματα ψηφοφορίας παρακαλώ να ψηφίσετε πιο γρήγορα πιέστε το κουμπί Πέρας. Εγκρίνεται. 24-13. Οπότε περνάμε. Τέσσερα πενήντα πέντε. Head. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άρθρο 11. Συμβαστική 73. Ποιοι είναι υπέρ. Α. Προφορικές τροπολογίες που ζήτησε το ECR, οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ. Έχετε στο κατάλογο σοφοριων σα. Έχει εγκριθεί από του σκιώδει. Ποιοι είναι υπέρ με την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφώ. Θέλει κανένα να ελέγξουμε, όχι, ωραία. Οπότε, περνάμε, περνάμε πολύ καλή συμβαστική προσπάθεια των εισηγητών αυτή. Οπότε περνάμε διάφορες σελίδες. 583 De Δεν θα την αποσύρει. Ψηφίζουμε. Κατά. Απορρίπτεται. 584 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 16 Συγγνώμη, 16. Συμβαστική 54. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 17. Έχουμε δύο ταυτόσιμες υπέρ κατά. Απορρίπτονται. 604 και 20 λέει ο, ο πρόεδρος. τώρα λέει 604 και 25 της απασχόλησης. Υπέρ. Ωραία. Με, μερικοί τα έχουν παρατήσει. Δεν ψηφίσουν καθόλου. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. Τρέχω τόσο πολύ. Δεν ήταν από κοινού. Πρέπει να ψηφίσουμε την Regi 37. Να επανέλθουμε σε αυτήν. Regi 37. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 604 απορρίφθηκε ηλεκτρονικά. Έμπλη 25. Υπέρ. Έμπλη 25. Θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία γι' αυτό. Πέρασε. Απορρίπτεται. 602 λοιπόν τώρα. 602 της κυρίας Ρούλε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστικές 55 και 52. Από κοινού, υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Οπότε, περνάμε στην 40, 41 κτλ. Αυτές θα ψηφιστούν από κοινού. Υπέρ. Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται, άρχεται για αυτές τις ε, από κοινού. Πέρας. Εγκρίνονται. Ήτρε 39, γιατί της κυρίας Βέσφαλ έχει αποσυρθεί υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 616 και τα λοιπά ταυτόσημες υπέρ. Λοιπόν, ηλεκτρονική. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας εγκρίνονται 21-18, 21-18 Ήτρε 40 άρχεται πέρας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά μία αποχή οπότε 6-18 με την προφορική τροπολογία ηλεκτρονική 618 συν προφορική. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ρέτζι 40 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 56 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 51 υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. 645-646, 45-46 ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τραν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία του κυρίου Ζουβά υπέρ κατά απορρίπτεται. Ίντα 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Οπότε τώρα περνάμε στη συμβαστική 3 υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε Λοιπόν, συμβαστική συμβαστική Κατά. Εγκρίνεται. 661. Ταραμπελά. Άρχεται για την 661. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για την 662. 662 υπέρ. Υπέρ. Όχι, όχι. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονική. Να ελέγξουμε. 662. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 664 από τον εισηγητή, τροπολογία. 664 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 666 της κυρίας Χάρκιν. 666 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Ρέτζι 41. 41 με συγχωρείτε. 41 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 669 Το κύριο Βαντεκάμπ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία αυτή. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο επιπλέον υπέρ. Σας παρακαλώ να πατάτε το κουμπί 670. Άρχεται η ψηφοφορία για την 670. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 671 της κυρίας Γκέπχαρτ Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 671. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στη συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα 670-671 Άρχεται η ψηφοφορία για αυτήν την αποκοινού ψήφιση. Ε, το ΕΛΚ εδώ έχουμε μία ψήφο παραπάνω. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 683 Διόν, Δε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορια απορρίπτεται 685 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Σαφώς τώρα περνάμε 48, 50 και 54 από τον εισήγητη, από κοινό ψηφοφορία των τριών τροπολογιών του εισήγητη. Σας παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται και οι τρεις απορρίφθηκαν. 691, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, απορρίπτεται. 693, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 693. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 692, 692 Άρχεται η ψηφοφορία για την 692 692 πέρας της ψηφοφορίας Ένα σήμα διαφορετικό μου ήρθε, γι' αυτό με συγχωρείτε. 694. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 695. Κύριε ε, Σβάμπ. Ναι. Ναι, ναι, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. Μετά έχουμε τροπολογίες που θα ψηφιστούν από κοινού, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ε, Ήτρε 45, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ, κατά, σαφώς εγκρίνεται. 703 της ε, κυρίας Χάρκιν απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική 7, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην ε, τροπολογία 709, ε, Ρέτζι, υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 52 του εισηγητή, υπέρ, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 708. 708 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 710 και Ρέτζι 146 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 711 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και ως προσθήκη 712 713 υπέρ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 7.14 υπέρ κατά απορρίπτεται. 7.15 υπέρ κατά απορρίπτεται επίση 7.16 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7.18 υπέρ, υπέρ, νομίζω καλύτερα ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε. 7.18 άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται 21 υπέρ, 17 κατά, 718, 719 καταπίπτει, 720 ψηφίζουμε, 721 καταπίπτει, 722, 722 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 726 726 άρχεται η ψηφοφορία για την 726. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 747 του εισηγητή υπέρ, κατά, Χρειάζεται να ελέγξουμε νομίζω ηλεκτρονικά για την 747. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 748 υπέρ κατά εγκρίνεται. 750 υπέρ 750 κύριε Σφάμπ 750 υπέρ υπέρ δεν είδα πολλά χέρια να σηκώνονται. Κατά. Απορρίπτεται. 751. Υπέρ. Κατά. Επίσης απορρίπτεται. 749. Καταπίπτει. Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε. 749 ψηφίζουμε. 749 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 46 υπέρ κατά απορρίπτεται 752. 752 πρέπει να ελέγξουμε για την 752. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά σε ελέγξουμε να είμαστε βέβαιοι. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 754 υπέρ. Και πάλι ας ελέγξουμε 754. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε 20 κατά 18 υπέρ. 755 Άρχεται η ψηφοφορία για την 755 πέρας της ψηφοφορία. Απορρίφθηκε επίσης. Ήτρε 47 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 55 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 756 αποσύρθηκε, κύριε Κρόιτσμαν. 757 Άρχεται η ψηφοφορία για την 757. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56 καταπίπτει. 758 της κυρίας Ρούλε υπέρ κατά απορρίπτεται 759 και 760 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. 761. Το 755 εγκρίθηκε. 761 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 764 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Reggie, 48 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 762 υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς 763 υπέρ κατά εγκρίνεται 765 ήδη καλύφθηκε από την Ρέτζη 48 απορρίφθηκε 766 υπέρ κατά απορρίπτεται Ήτρε 48, πρόκειται για γλωσσική τροπολογία, 767, 768 υπέρ, εγκρίνονται. Ήτρε 49, υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Ηλεκτρονικά. Μικρή πλειοψηφία, νομίζω. 22 υπέρ, 15 κατά, 769 υπέρ, υπέρ, κατά. δεν είναι σαφή τα πράγματα, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αν μπορείτε σαφέστερα να σηκώνετε τα χέρια σας για να μπορούμε να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Ναι, δεν μπορούσα να κρίνω χωρίς ηλεκτρονικό έλεγχο. 770 υπέρ, υπέρ, παρακαλώ σηκώστε τα χέρια. Θα πρέπει να ελέγξουμε, με συγχωρείτε. Πέρα της ψηφοφορίας, 21 κατά, 17 υπέρ, 771 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 57 καταπίπτει. 772. Α, θα ψηφίσουμε για την 57 ως προσθήκη. Επανερχόμαστε λοιπόν στην 55 του εισηγητή. Με συγχωρείτε. 57 ως προσθήκη. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7-7-2. 772. Άρχεται η ψηφοφορία για την 772. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 773, 774 καλύφθηκαν. Ρέτζι 49. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται, σαφώς. 775 αποσύρθηκε, 776 776 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Περνάμε στις συμβιβαστικές 11 και 12 υπέρ κατά εγκρίνονται σαφώς και τώρα περνάμε στην 814 υπέρ κατά απορρίπτεται 8-15 ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ρέτζι 52 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 8-17, 8-18 από κοινού, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 8-16 ως προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 8-19 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 8-20 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 8-21 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 43 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην ε, συμβιβαστική 44 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 45 συμβιβαστική υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 862, 862 τροπολογία Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για την τροπολογία 862. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ήτρε 54. Ήτρε 54. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Right, Yeah. Ναι, ναι. Κατα... Ε, απορρίπτεται. 863. 863 υπέρ, κατά, απορρίπτεται σαφώς. MV30 που απορρίπτεται επίσης. Συμβιβαστική 46 υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Και τώρα περνάμε στην ε, τροπολογία 870 της κυρίας Ρούλε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 871 υπέρ, και πάλι εγκρίνεται. 872 υπέρ. Θα πρέπει να ελέγξουμε. 872. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 873. 873. Ναι. Θα ελέγξουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης 874, ε, 875 υπέρ, κατά, απορρίπτονται 876 ε, από κοινού μέχρι το, την 882 από κοινού όλες αυτές οι τροπολογίες υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 879 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ρέτζι 55 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 881 της κυρίας Ρούλε υπέρ, κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Εντάξει. πέρα στις ψηφοφορια Απορρίπτεται. 20 κατά 17 υπέρ, 883 της κυρίας Χάνσλικ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 884 της κυρίας Χάνσλικ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 885 της κυρίας Χάνσλικ υπέρ κατά επίσης απορρίπτεται. Συμβιβαστική 57 υπέρ κατά εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά εγκρίνεται. 20 συμβιβαστική, 28 συμβιβαστική τροπολογία 28. Καλά πάμε. Για το άρθρο 41. Υπέρ, Α, είναι χωριστή η ψηφοφορία, μάλιστα. Συμβιβαστική τροπολογία 28. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με σαφήνεια. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Και αυτό εγκρίνεται σαφώς. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Και αυτό εγκρίνεται. Περνούμε λοιπόν στη συμβιβαστική τροπολογία 29 29. Ναι. Πολύ σωστά. Δεν χρησιμοποιώ τις σελίδες γιατί τα κινη... Άρθρο 42. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Συμβιβαστική τροπολογία 50. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Στη συνέχεια άρθρο 989. Α, έχει αποσυρθεί. Οπότε συμβιβαστική τροπολογία 41. Υπέρ, κατά. Και αυτό εγκρίνεται σαφώς. Περνούμε λοιπόν στην 62 Επιτροπή Περιφερειό για τα περιφερειακά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Α, απορρίπτεται αυτή. 63 Ρέτζι. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Επομένως η 6 καταπίπτει. Υπάρχει μια προσθήκη. Ας ψηφίσουμε. Πιστεύω ότι θα απορριφθεί ούτως ή άλλως, αλλά υπέρ, κατά, χάνουμε το χρόνο μας εδώ πέρα, τέλος πάντων. Επιτροπή Βιομηχανίας. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1-1-9. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θέλω και ένα σήμα από την πλευρά σου, Ντένις, να μου δείχνεις καθαρά. 1, 1, 0, 9. Παρακαλώ λίγο πιο γρήγορα να πατάτε τα κουμπιά. 34 φτάσαμε εκεί. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 21, 15. 1-0-2-1. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 25 γιούρι υπέρ κατά, απορρίπτεται. 1-2-2 υπέρ, κατά, απορρίπτεται επίσης. 1-0-4 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 105 Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1.06. Όχι. 1.07. Υπέρ. Κατά. Μάλλον χρειαζόμαστε έλεγχο. Ας ελέγξουμε. Η πλειοψηφία δεν είναι σαφής. Εγκρίνεται. Η 107 εγκρίθηκε. Γιούρι 26 υπέρ. Α, με συγχωρείτε. 102.8. 102.8 υπέρ. 1.028 υπέρ. Ε, απορρίπτεται. Τζούρι 26. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στο άρθρο 73, 1022, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1458, τροπολογία υπέρ, κατά, και αυτή απορρίφθηκε. 1459, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1-4-1 του εισηγητή, υπέρ, κατά, επίσης απορρίφθηκε. Α, όχι, αυτό δεν το έφερε. Εντάξει. Συμβιβαστική τροπολογία 30 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ, 31, σελίδα 75, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περάσαμε τη σελίδα 75 από τις 150. Έχουμε κάνει τα μισά λοιπόν. Α, φτάσαμε στην σελίδα 80. Έχουμε περάσει λοιπόν σαφώς το δεύτερο μέρος. Συμβιβαστική τροπολογία 32. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 1093 υπέρ κατά Δεν είδα τι έκαναν οι πράσινοι, επομένως θα ελέγξουμε. Α, αποχή! Ας ψηφίσουμε τότε. 1093, ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται περνούμε στην 102-103 ε, του εισηγητή μαζί, υπέρ. Αρχή της ψηφοφορίας, πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο, με μία ψήφο. 1094 υπέρ. Απορρίπτεται. 1095. Υπέρ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 1095. Ε, Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 13 κατά. 1096 της κυρίας Χάνσλικ. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 1097 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 105-46 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά απορρίπτεται. Υπάρχουν αποχές. Απορρίπτεται. 1098 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1099 υπέρ κατά απορρίπτεται. 106 του εισηγητή Νομίζω ότι θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 106 του εισηγητή. Πέρα της ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας. Κάποιος άλλαξε τη γνώμη. Κάποιος άλλαξε γνώμη. Ο κύριος Σβάμπ άλλαξε τη γνώμη του μόλις κοίταξε την οθόνη. Συμβιβαστική τροπολογία 39. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνούμε τώρα στην 1106. 1106, ποιοι είναι υπέρ. 1106. Κατά, απορρίπτεται. Μετά 25 πεταφορών, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 107 και 47, ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχέ, ε, απορρίπτεται, 1107 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 108 υπέρ. Θα ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας, απορρίπτεται. 20 κατά 18 υπέρ. Απασχόληση 40 Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 1108 καταπίπτει. 1109 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 48 δεν τη βάζουμε. Τετραπλή. 1111. <laughs> 1-1-1-1. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1110. Υπέρ. Κατά. Αυτή εγκρίθηκε. 1113 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 110 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Παρακαλώ να μου να δείχνετε πιο έντονα. Απορρίπτεται. 1114, 1114 υπέρ, κατά, και αυτη απορριφθηκε 111. 1-1-1, 111 και 115. Αρχίζει η ψηφοφορία. πέρασε τη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Με δύο μόνο ψήφους. All right. So we can still add the words. So, so no, no, we vote the whole amendment 1116 and 14. All right. So we, we vote. Ψηφίζουμε την 1116 ε, ως προσθήκη. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Φιλελεύθεροι, μπορείτε έτσι πιο δραστήρια να μου δείχνετε τι ψηφίζετε. Πιο εμφατικά, παρακαλώ. 82. Βιομηχανίας. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Νομικών υποθέσεων 32. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τζούρι 33. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1117 και 83. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 1118 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 1119 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 113 υπέρ, έλεγχος, ελέγχουμε για την 113 1-1-3 του εισηγητή. 1-1-3. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 1-1-2-0 του εισηγητή υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 72 περιφερειών ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 120... Δεν τη βάζουμε αυτή. Συμβιβαστική τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, ναι. Κυρία Κοράτσα Μπίλντ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ψηφίσουμε χωριστά την 1165 στη σελίδα 89 να την ψηφίσουμε ως προσθήκη, γιατί καλύπτεται και αυτή από τη συμβιβαστική τροπολογία 33. Κριτήρια σύμβασης, ε, ε, κριτήρια κόστους ωφέλειας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ταραμπέλα και τον σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ που το στήριξε και ελπίζω και οι άλλοι να μπορέσουν να στηρίξουν. Ε, είναι προσθήκη στην λίστα ψηφοφορίας του ΕΛΚ. Εάν συμφωνεί ο εισηγητής, εντάξει, θα το αφαιρέσω από τη συμβιβαστική τροπολογία και θα το ψηφίσουμε χωριστά. Δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν έχει και κανείς άλλος αντίρρηση. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε πάνω στην συμβιβαστική τροπολογία ως έχει, 33. Μετά οι προσθήκες υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Κρίνεται σαφώς. Οπότε τώρα πηγαίνουμε στην 1165 ως προσθήκη. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και αυτό. Οπότε τώρα περνούμε κατευθείαν στη συμβιβαστική τροπολογία 34. Σε δύο τμήματα η ψηφοφορία. 34 τμήμα 1. Υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ, κατά και αυτό εγκρίνεται. Περνούμε τώρα 1, 2, 3, 4 από κοινού 1, 2, 3, 4 και τα Συγγνώμη, 1243 ε, διορθώνει ο πρόεδρος.

υπέρ, κατά, απορρίπτονται όλες. Συμβιβαστική τροπολογία 35, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επομένως, περνούμε μετά απευθείας στο άρθρο 70. Τροπολογία 1304 του κυρίου Σφάμπ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνούμε λοιπόν στις... στη 1315 και 16. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται αυτές. Ρέτζι 81 και 1317 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 153 του εισηγητή υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Περιβάλλοντος 69 και 61. Α, δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Και μετά από κοινού 94 έως 97. Υπέρ, κατά, όλες απορρίφθηκαν. 1318 και 1319. Υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, ε, απορρίπτονται. Συμβιβαστική τροπολογία 37. Σε έξι τμήματα. Χωριστή ψηφοφορία σε έξι τμήματα. Τμήμα 1 και 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τμήμα 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τμήμα 4 υπέρ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, εντάξει. Αρχίζει η ψηφοφορία για το τμήμα 4. Θα ελέγξουμε, θα ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Εγώ το, θα το έλεγα, το είχα καταλάβει. Αλλά είναι καλό να γίνεται έλεγχος. Καταπίπτει το τμήμα 5 λοιπόν. Ψηφίζουμε το τμήμα 6. Όχι, δεν εγκρίθηκε. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Τμήμα 5 ψηφίζεται τελικά. Υπέρ για το τμήμα 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Και τμήμα 6. Υπέρ. Κατά. Και αυτό εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν περνούμε στη συμβιβαστική τροπολογία 58 υπέρ Α, σε τρία τμήματα, μάλιστα. 58. Ξέρετε πόσο μας αρέσουν εδώ οι ε, χωριστές ψηφοφορίες. Κάποιος τρίζει τα δόντια του. Συμβιβαστική τροπολογία 58 τμήμα 1. Υπέρ. Κατά αυτό εγκρίθηκε. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Και αυτό εγκρίνεται. Τμήμα 3. Υπέρ. Κατά. Και αυτό εγκρίθηκε. Όλα εγκρίθηκαν. Συμβιβαστική τροπολογία 47 η οποία επίσης χωριστεί ψηφοφορία, με μια προφορική ε, τροπολογία από το ECR. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Περνάμε στην 1386. Υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. Χίλια υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Ε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Περνούμε τώρα στην 75, 76 και 77 από κοινού, αλλά με χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Τμήμα 1, όπως φαίνεται στη λίστα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τμήμα 2, υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Τμήμα 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται επίσης. Περνούμε τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία 79. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνούμε στη συμβιβαστική τροπολογία 71. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 1396 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1431 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 50 απασχόλησης υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1443. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1444 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 103 βιομηχανίες υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. 59. Συμβιβαστική τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 60. 60. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν περνούμε στην 110 της Επιτροπής Βιομηχανίας υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 61 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 1523, 1523 και τα λοιπά. Όλα είναι διαγραφές. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 62. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 1528. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1530. Απορρίπτεται. 1544 έφυγε, 1545-46 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συμβιβαστική τροπολογία 63. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία... Συμβιβαστική τροπολογία 64. Υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. Είναι τα 41, τραν 45. Υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Είναι τα 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ήτρε 112 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ήτρε 113 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, είχε ήδη απορριφθεί, επειδή απορρίφθηκε 112. 1560 ρούλε υπέρ. <clears throat> Κατά. <clears throat> Χρειάζεται να το ελέγξουμε. 1560. <clears throat> Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 78. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Κατά τμήματα. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα της συμβαστικής 27 υπέρ. Κατά εγκρίνεται σαφώς. Και το δεύτερο τώρα της 27 πάντα συμβαστικής υπέρ λοιπόν. Υπέρ. Ωραία, θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 27. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε, οπότε, είναι τα 43 και τα λοιπά, παράρτημα 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Άλλο ένα μπλοκ ψηφοφοριών, Σαλβίνη και Σπερώνη, που δεν, ε, δεν ξέρω ποιος ψηφίζει για τον κύριο Σαλβίνη σήμερα υπέρ κατά απορρίπτονται συμβαστική 40 υπέρ κατά εγκρίνεται οπότε οπότε 1581 πρέντακαστ υπέρ κατά απορρίπτεται 50-80 υπέρ κατα 1580. συγγνώμη υπέρ κατά απορρίπτεται 165 και τραν 46 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 1583 υπέρ. Υπέρ, υπέρ. Έλεγχος. 1583 μπέλετ. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 1582 παρακαλώ τώρα. 1582 υπέρ κατά απορρίπτεται 166 του εισηγητή υπέρ κατά απορρίπτεται απορρίπτεται 168 head υπέρ έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος για την αμφίροπο. Πέρας. Απορρίπτεται. 167 παρακαλώ. 167. Ηλεκτρονικά. 167. Νομίζω θα έχουμε τον ίδιο συσχετισμό αλλά μήπως ε, άλλαξε κανείς άποψη. 167 πέρας απορρίπτεται επίσης. Συμβαστική 81 υπέρ κατά εγκρίνεται. 171 υπέρ να ελέγξουμε 171 παρακαλώ. Άρχεται 171. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 82 υπέρ. Υπέρ. Χρειάζεται έλεγχος επί της συμβαστικής 82. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά, λοιπόν. Εμπλ 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ένβι 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1 Τροπολογία 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ρέτζι 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 175. Πίτι Κάινεν. Υπέρ. 175 λέγω. Κατά. Απορρίπτεται. NV1. Υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε MV1 παρακαλώ έλεγχος πέρας απορρίπτεται είναι τα υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς 174. Κοράτσα Μπίλτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην ίντα 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 177 και NV 3. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 180. Υπέρ κατά απορρίπτεται 179 υπέρ κατά εγκρίνεται MV5 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 84 υπέρ υπέρ πρέπει να ψηφίσουμε συμβαστική 84 άρχεται πέρας απορρίπτεται δύο ψήφοι διαφορά. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε μία-μία τις τροπολογίες τώρα. 181 και NV14. NV4. Υπέρ κατά. Απορρίπτονται. Έμπλ 3. Το αντίστοιχο τμήμα. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία από αυτού. Έμπλ 3. Το αντίστοιχο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. 186. Υπέρ. Υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να την ψηφίσουμε. Την 186. Πέρασε. Εγκρίνεται. Οπότε όλες οι άλλες καταπίπτουν. Οπότε περνάμε Έμπλ 4. Η Έμπλ 4 δεν καλύπτεται. Χρειάζεται να ψηφίσουμε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται υπέρ κατά απορρίπτεται όχι 188 λοιπόν και Ρέτζι 13 Ρέτζι 3 υπέρ κατά απορρίπτεται Απορρίπτονται MV7 υπέρ κατά απορρίπτεται Ήτρε 4 και NV8 υπέρ κατά απορρίπτονται 190 υπέρ κατά απορρίπτεται 4 του συγητή άρχεται πέρας απορρίπτεται Ρέτζι 5 λοιπόν ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται Ήτρε 5 υπέρ Υπέρ. Κατά. Σαφώς απορρίπτεται. Ίντα. 3, 4 και 5 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Ήτρα 6. Και εισηγητής 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Ίντα 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 195 υπέρ κατά απορρίπτεται. 197 κλπ. Όλες μαζί υπέρ κατά εγκρίνεται. Όλες αυτές εγκρίνονται. Συμβαστική 86 υπέρ, γιατί άλλες καταπληκτούν υπέρ. 86, 86 παρακαλώ υπέρ, κατά εγκρίνεται. Στην αιτιολογική σκέψη 13 έχουμε ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Ήτρο 8 ως προστίκη, υπέρ. Υπέρ λοιπόν, κατά. Απορρίπτεται. 209, ρούλε, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 87, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 2.15 2.15 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά επειδή είναι δική μου η τροπολογία ας ελέγξουμε για να μην νομίζετε ότι Και όντως εγκρίνεται 21 με 16. Τροπολογία 2.16 Ζουβά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε τροπολογία, τροπολογία 2.2.2 και 2.24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 2.23 Α, όχι, δεν ψηφίζουμε 2.23. Ψηφίζουμε 2.25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.26. Όχι, δεν την ψηφίσουμε. Λοιπόν, συμβαστική 88. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.31 υπέρ κατά κατά παρακαλώ ε, όσοι είναι κατά αποχές ψηφίσανε οι φιλελεύθεροι όχι 2.31 2.31 τροπολογία 2.31 σας παρακαλώ ψηφίστε έλεγχος Δεν ήταν σαφές. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 89 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 2.34. Μόνο αυτές τις λέξεις. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.35 υπέρ κατά εγκρίνεται 2.36 υπέρ κατά εγκρίνεται Α, όχι, να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε καλύτερα. 2.36. Κοράτσα μπίλτα. Δεν ήταν απόλυτα σαφές. Πέρασε. Εγκρίνεται 20-14. Τροπολογία 11 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 48. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 25. Οι τροπολογίε 241-242. Ε, Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.44. Μα μόλις ψηφίσαμε τις 2.41, 2.42. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Υπερβάλλω. Εγκρίναμε τη 49. Οπότε είμαστε τώρα στη 41-42. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Πάμε λίγο παραπίσω. Συμβαστική 49 υπέρ κατά εγκρίνεται 2.41 2.42 ταυτόσιμες υπέρ κατά σαφής απόρριψη σαφής έγκριση Ωραία, είναι σαφές. 2.44 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ρέτζι 6 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ κατά σαφώς απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 14 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα το δεύτερο υπέρ κατά επίσης εγκρίνεται. Οπότε ήτρε 14 υπέρ κατά απορρίπτεται. 250 υπέρ υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεν συμφωνεί ο κύριος Φάμπ Σκιώδης, αλλά εγκρίθηκε παρόλα αυτά. Έμπλ 10 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 17 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 42 υπέρ Κατά εγκρίνεται σαφώς. Αιτιολογική σκέψη 30. Κοράτσα Μπίλτ. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Ρέτζι 8. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 53. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Και μετά έχουμε ε, μαζί 15, 16, 19, 20 ήτρε υπέρ. Απορρίπτονται. Ήτρε 21. Α, ήταν με στο μπλοκ. Πάει. 2.55 και έμπλ 11. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Ήτρε 22 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 18 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 270 υπέρ κατά εγκρίνεται 271 Θέλετε να κάνετε προφορική τροπολόγηση της τροπολογίας σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφορική στη 271 για την αιτιολογική σκέψη 38β. Για το θέμα αυτό η αρχή που συνάπτει το συμβόλαιο μπορεί να λάβει υπόψη τις μεθόδους παραγωγής και, και για την ε, ε, διατύπωση των ε, κριτηρίων αξιολόγησης με πλήρη συμμόρφωση με τον κοινοτικό νόμο. Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές συμφώνησαν νομίζω ότι θα είναι συν για το ΕΛΚ εάν εγκριθεί αυτή η προφορική συμπλήρωση. Ωραία, ας το ψηφίσουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Ωραία, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 του εισηγητή υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 272. Όχι. Όχι. 272 υπέρ κατά απορρίπτεται. MV15 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 24 ως προσθήκη υπέρ κατά όχι, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ως προσθήκη. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, Ήτρε 26 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2,78 και 2,79 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Συμβιβαστική 21 σε τμήματα χωριστά. Ψηφίζουμε για το τμήμα 1 υπέρ, υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς. Τμήμα 2 υπέρ θα ελέγξουμε για το τμήμα 2. Τμήμα 2 για τη συμβιβαστική 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους ε, υπέρ ε, επιπλέον των κατά. 20 υπέρ, 17, 22 ε, εγκρίνεται. 23 κατά εγκρίνεται. 297 γκρέκα υπέρ, υπέρ, κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. «2.97» άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 2.97. πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 21 υπέρ 16 κατά 2.98 δεν ψηφίζουμε ούτε για την Τζούρι 7. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά εγκρίνεται λογική σκέψη 47, έμπλ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 302 και άλλες υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 303 της κυρίας Ρούλε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται, συμβιβαστική 91, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 301 υπέρ, όχι, όχι. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, προχώρησα πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος. Είστε στην τελευταία σελίδα τώρα. Δεν υπάρχουν άλλες πρόσθετες σελίδες. Συμβιβαστική 92, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Σαφώς 311 ε, ε, υπέρ, κατά, θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 311. ...311. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 22 του εισηγητή υπέρ κατά απορρίπτεται. Ρέτζι 15 15 υπέρ κατά απορρίπτεται επίσης. Τροπολογία 312 υπέρ κατά εγκρίνεται. 313 υπέρ κατά. Δεν ξέρω για να δούμε το αποτέλεσμα, να ελέγξουμε, είναι αμφίβολο, 313 Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 20 υπέρ 18 κατά. Αυτό σημαίνει ότι η 314 καταπίπτει. Περνάμε ε, στην τραν 1. Όχι. Ρέτζι 16, με συγχωρείτε. Ρέτζι 16 υπέρ. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την Ρέτζι 16. Yeah. That's carried. Εγκρίνεται. Ρέτζι 17. Ρέτζι 17. Υπέρ. Ρέτζι 17. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 317 της κυρίας Ρούλε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 318 του κυρίου Ντεγιόγκ. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. τα 15 υπέρ κατά απορρίπτεται. 3.20 υπέρ κατά Δεν μπορώ να δω καλά. Δεν μπορώ να δω καλά. Ας ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Right. 321 και 22 Ρούλε και Ντε Ιόγκ υπέρ κατά Α, και πάλι δεν αμφιβάλλω. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, είναι η τελευταία ψηφοφορία. Τελευταία. 20 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Πολύ καλά. Τώρα έχουμε την τελευταία ε, γνωμοδότηση, αν θέλετε, της Επιτροπής που ψηφίζεται. Ανοιχτή ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 8 κατά και 7 αποχές. Εγκρίθηκε η γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Τελειώσαμε για σήμερα το πρωί. Uh, πρωτού φύγουμε από την αίθουσα. Παρακαλώ ησυχία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο εισηγητής θέλει να προσθέσει κάτι ε, προτού λύσουμε τη συνεδρίαση μέχρι το απόγευμα. Θέλετε το λόγο, όχι. Θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπα προηγουμένως, ευχαριστώντας άλλη μια φορά τη γραμματεία σας, εσάς προσωπικά, τον πρόεδρο, αλλά ακόμα και τους σκιώδεις συγητές για την εργασία η οποία έγινε. Βεβαίως θα πρέπει να μελετήσουμε το σύνολο των ψηφοφοριών για να δούμε αν το μήνυμα είναι σαφές, να δούμε όλους τις συμβιβασμούς, το σύνολο των συμβαστικών ε, τροπολογιών εγκρίθηκαν εκτός από δύο στις αιτιολογικές σκέψεις. Δεν ήταν λοιπόν άχρηστο να δουλέψουμε μαζί, να συνεδριάσουμε, να ξανασυνεδριάσουμε, να ανταλλάξουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Το μήνυμα είναι σαφές, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα κείμενα, ούτω ώστε να δούμε αν δεν υπάρχει αντίφαση ανάλογα με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Οι συμβιβασμοί ήταν πολυπληθείς, πολυπληθείς και βεβαίως έτσι δεν δίρκεσε όλο το πρωινό η ψηφοφορία και τώρα μπορούμε να ξεδιαλύνουμε την θέση του Κοινοβουλίου. Θα τελειοποιήσουμε την θέση αυτή, θα απέναντι και στο Συμβούλιο που εργάστηκε παράλληλα πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε μια θέση και ένα σαφές μήνυμα ήταν ο στόχος που θέλαμε για αυτό το θέμα που ήταν περίπλοκο και αυτή, ήταν η, αυτή είναι η ουσία του μηνύματος που θέλουμε να μεταδώσουμε. Θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα απλά, να πάρουμε τους κατώτερους κανόνες και τα πράγματα θα ήταν απλά, αλλά θέλαμε να δώσουμε εργαλεία στις αναθέτουσες αρχές για να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα κονδύλια στις επενδύσεις σε εργασίες, σε αγαθά, σε υπηρεσίες και να μεριμνήσουμε ούτω ώστε οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές να μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα σε όλο το πλαίσιο ε, των δημοσίων συμβάσεων. Θα υπάρχει το Συμβούλιο, η Κομισιόν που είναι ένας εταίρος που αρχικά είχε ένα έγγραφο προς τη σωστή κατεύθυνση και μας βοήθησε πάρα πολύ και τώρα κλείνω ευχαριστώντας για το εξαίρετο πνεύμα συνεργασίες που υπερήχε για το θέμα αυτό, διότι κανένα από τα μέρη δεν έχει την πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο, γι' αυτό πρέπει πάντοτε να επιζητούμε συμβιβασμούς. Εμείς οι Βέλγοι το ξέρουμε καλύτερα λόγω της χώρας μας. Ήταν μεγάλη χαρά που εργαστήκαμε για αυτό το θέμα το περίπλοκο, αλλά που είναι σημαντικό για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης και για το μέλλον των δημοσίων δαπανών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων την ομάδα που συνέταξε τον κατάλογο ψηφοφοριών διότι το γεγονός ότι τελειώσαμε περίπου μια ώρα νωρίτερα, αυτό οφείλεται στην προετοιμασία του καταλόγου των ψηφοφοριών. Ξέρω ότι χρειάστηκε να δουλέψουν πάρα πολύ, πολύ αργά για να γίνει αυτός ο κατάλογος ψηφοφοριών. Θα ήθελα να σας πω ότι τελειώνουμε πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, αλλά ε, πρέπει να αρχίσουμε στις 3 ε, το απόγευμα. Θα επανέλθουμε εδώ στις 3 το απόγευμα. Ίσως μπορέσουμε... Μετά έχουμε την ε, εισήγηση του κυρίου Ραμών θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε την Κομισιόν παρούσα για την έκθεσή του και θέλετε να νομίζω να αρχίσουμε νωρίς, να τελειώσουμε όλοι νωρίτερα, να είστε εδώ στην ώρα σας. Θα υπάρχει επίσης ένα, μια άτυπη συνάντηση με τον τύπο και ο εισηγητής και οι σκιώδης θα ε, συμμετάσχουν. Θα γίνει εδώ αυτή η συνάντηση Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο Press Point, ε, ας μην έρθουν. Ε, τώρα κλείνουμε τη συνεδρίαση και θα ξαναβρεθούμε εδώ στις 3. And our interpreters are going to stay to help us with the press as well, I think.